Πριν ε, κηρύξω την άνοιξη συνεδρίασης, κύριε και κύριοι, θα ήθελα να κάνω επανάληψη να σα επισημάνω την περασμένη εβδομάδα ε, από τρομακτικά, ε, τρομοκρατικά χτυπήματα του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους για τις επιθέσεις στην Τουρκία, στην Ιαμένη, στον στο και στο Ιράκ ε, οι τόποι αυτοί εντός ε, ολίγων ημερών στόπους αυτούς ε, σκοτώθηκαν 300 άτομα και πληγώθηκαν 400. Μεταξύ των θυμάτων άνδρες και γυναίκες, πολλά παιδιά, ενοπλοί και άμαχοι, άνθρωποι διαφόρων προελεύσεων με διαφόρων θρησκευμάτων και εθνικοτήτων. Η διεθνής Ρωμοκρατία αυτής της ομάδας πραγματικά δεν κάνει διακρίσεις στα θύματα ε, και προσβάλλει και πλήττει τους πάντες. Ο Πρωθυπουργό ε, του Μπασουλαντές, ο Σέικ Χαζίνα, είπε πολύ ορθά ότι αυτή η τρομοκρατία, αυτή η μορφή τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα και δεν γνωρίζει θρησκεύματα. Καταδικάζουμε αυτές τις ε, γεμάτο, γεμάτες μίσος επιθέσεις ε, σενάρα και είμαστε ενωμένοι με τους άλλους λαούς έναντι μια τέτοιας απειλής την οποία θα πρέπει να καταπολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και προωθώντας την υπεράσπιση των δικών μας αρχών. Ε, κανένας πολιτικός στόχος δεν δικαιολογεί την ε, χρήση αυτής θερατόδους βίας. Αυτή η δημοκρατία χωρίς σύνορα και αυτή η φωνική ιδεολογία μπορεί να καταπολεμηθούν μόνο μέσω μιας στρατηγικής ε, παγκόσμιας συνεργασίας. Όλοι βρισκόμαστε βεβαίως σε πένθος και θα ήθελα να πω στις οικογένειες των θυμάτων και στους, ε, στους οικείους και ε, στις χώρες ε, τους τα συλληπιτήριά μας και θα ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα αυτά. Τα πρακτικά και τη συνεδρίαση τη 26η και 27η, καθώ και τα πρακτικά τη έκτατη συνεδρίαση τη 25η Ιουνίου και στις